έγκυρες θητείες του κυρίου Ντανιέλ Ντάλτον από την 8 ε, Ιανουαρίου 2015, την εντολή του κυρίου Στέλιου Κούλογλου από τις 27 Ιανουαρίου 2015, την εντολή της κυρίας Ανελίν Βαν Μπόσοιτ 8 Ιανουαρίου 2015 και Χίλντε Βάουτμανς 1 Ιανουαρίου 2015. Προτείνω να εγκρίνουμε αυτές τις εντολές των συναδέλφων. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε και εγκρίνονται και οι τέσσερις αυτές εντολές.